Πριν περάσουμε στις ψηφοφορίες, έχω μία δήλωση να ε, διαβάσω. Θα θυμάστε ότι ο πρόεδρος κατά τη συνεδρίαση στις 11 Μαΐου 16 επέβαλε μία κύρωση στο συνάδελφο Συναδεινό γιατί έκανε απαράδεκτες ε, δηλώσεις για τον τουρκικό πληθυσμό κατά την Ολομέλεια της 9 Μαρτίου. Στο Προεδρείο τη Δευτέρα 6 Ιουνίου με την ένσταση του κυρίου Συναδεινού και ομόφωνα αποφασίσαμε να βεβαιώσουμε την απόφαση του Προέδρου. Η κύρωση είναι η αφαίρεση 10 ημερήσεων ε, αποζημιώσεων από τον κύριο Συναδεινό και πληροφορήθηκε γι' αυτό χθε. Να περάσουμε τώρα στις ψηφοφορίες.